Okay. Okay. Um... Λοιπόν, ε, ξεκινάμε την ε, συνεδρία της Επιτροπής. Μόλις έχουμε καταφέρει να έχουμε αρκετούς βουλευτές για να μιλήσουμε για τα διάφορα θέματα. Πρώτα απ' όλα έχουμε το σχέδιο μέσης διάταξης. Ζητήθηκε να υπάρξει αμοιβαία ανταλλαγή των δύο πρώτων ψηφοφοριών και αν δεν έχει κανείς καμιά αντίρρηση θα το κάνουμε έτσι. Γιατί όλοι έχετε κάποια αεροπλάνα να προλάβετε. <coughs> Κάνω πρώτα τις ανακοινώσεις της Προέδρου. Ελπίζω να μην είναι τόσο λίγοι οι παριστάμενοι και να έρθουν και άλλοι. Πάμε στη συνέχεια, δεν έχω να πω τίποτα. Πάμε στο σημείο 3 που είναι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για το συντονισμό της Ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής με εισαγωγή τον Φίλιπ Τεμπάκερ και έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους για την πολύ καλή συνεργασία τους. Ξέρουμε ότι μερικές φορές αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερα επίμαχο, αλλά έχουμε εξετάσει όλες τις τροπολογίες, τις έχουμε μελετήσει, κάναμε μια καλή συζήτηση και τελικά καταλήξαμε σε κάποιες ε, ε, κάποιες συμβαστικές λύσεις που είναι πια αποδεκτές. Το μήνυμα είναι, εν πάση περιπτώσει, ότι η ετήσια οικονομική επισκόπηση θα πρέπει να λάβει υπόψη το γενικό πλαίσιο για την οικονομική διακυβέρνηση που έχει δημιουργήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα. Έχουμε δώσει μεγάλη σημασία στη συνέχιση των διαφορετικών μεταρρυθμίσεων. Επίση, είχαμε πολλέ ε, συζητήσει για το πώ θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα πιο ευνοϊκό κλίμα ανάπτυξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι και αντικείμενο μιας χωριστής έκθεσης και φυσικά το θέμα της Ταπεζικής Ένωσης και της περάτωσης, της αποπεράτωσης της Νομισματικής Ένωσης στην Ευρώπη είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει όλους και είναι μια μεγάλη προτεραιότητα. Είχαμε επίση και ένα κεφάλαιο για τη δημοκρατική λογοδοσία για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και εκεί συμφωνούμε ότι είναι πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν ακόμα. Νομίζω τελικά ότι και στον τομέα αυτό έχουμε διατυπώσει δύο καλές παραγράφους είναι λοιπόν πολύ εξισορροπημένη αυτή η έκθεση και ευχαριστώ όλους τους και όλους για τη συνεργασία τους και ελπίζω και στην ψηφοφορία ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια ευρία πλειοψηφία για αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον εισηγητή για το έργο που έχει φέρει σε πέρα στην έκθεση αυτή φαινόταν ότι ήταν πολύ δύσκολο το έργο του, αλλά χάρη στην καλή θέλησή του μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε να διεκπαιρεώσουμε αυτή την έκθεση χωρίς προβλήματα. Νομίζω ότι έχει καταφέρει μια εξισορροπημένη έκθεση, η οποία χωρίς καμία αφιβολία μπορεί να επιτύχει τον αρχικό στόχο που επιζητούσαν όλες οι πολιτικές ομάδες. Θα ήθελα να τονίσω ορισμένα ε, σημεία της ε, έκθεσης που <clears throat> καταγράφουν και εξέρουν τα διάφορα επιτεύγματα που έχουν γίνει και σε επίπεδο εθνικό και σε επίπεδο ευρωπαϊκό, τις πρόοδους λοιπόν που έχουν επιτευχθεί σε ό,τι αφορά την ε, οικονομική ολοκλήρωση, την Τραπεζική Ένωση, το ρόλο της Τράπεζας Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Η αρχική έκταση μας παρουσίασε <clears throat> ο εισηγητής περιείχε ήδη τις περισσότερες προτεραιότητες που η δική μου ομάδα ήθελε να εισαγάγει, επομένως δεν υπήρχε μεγάλους λόγους για τροπολογίες. Απλώς αυτό το οποίο θέλησαμε να κάνουμε είναι να τονίσουμε λίγο περισσότερο τον ε, ρόλο που πρέπει να έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην οικονομική ανάκαμψη και να υπογραμμίσουμε ότι στην τωρινή συγκυρία αυτές οι επιχειρήσεις, ιδίως αυτές που βρίσκονται στη ζώνη του ευρώ έχουν ιδιαίτερες δυσκολίες πρόσβασης σε χρηματοδότηση και επιστώσεις και πιστεύουμε ότι εδώ πρέπει να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να εξασφαλίσει ότι οι πιστώσεις θα γίνονται σε αντίστοιχες συνθήκες σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανεξάρτητα από την χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένη πάντα μέσα στη ζώνη του ευρώ. Επομένω, να γίνεται η επιλογή όχι από τη βάση γεωγραφική του θέση, αλλά επί τη βάση τη οικονομική του ε, ευρωστία. Λέω και πάλι ότι θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον εισηγητή και όλου όλε κοιόδη εισηγητέ, γιατί χάρη στην καλή του προσπάθεια ήταν εύκολο σχετικά το έργο μα και με ένα αποτέλεσμα το οποίο θέλω να περιγράψω ω ιδιαίτερα θετικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχουμε κάποιον σκιώδη εισηγητή από τους σοσιαλδημοκράτες εδώ, άρα περνάμε στον Τερκ Έπινγκ. Μιλώ εκ μέρους των συντηρητικών. Βλέπω ότι δεν υπάρχει και σκιώδη εισηγητής από τους φιλελεύθερους, εκτός από εσάς. Ναι. Είμαι, εισηγη... Ε, είμαι πρόεδρος, λέει πρόεδρος από τους φιλελεύθερους. Ξέρω πως είστε μακριά μου και δεν με βλέπετε. Θα βάλω τα γυαλιά μου λοιπόν, λέει ο κύριο Σέπινγκ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κύριο Ντεπάκερ, για την επικοδομητική και καλή δουλειά που έκανε στην έκθεση αυτή. Απέδειξε πω είναι ένα πάρα πολύ καλό εισηγητή, προσπάθησε να συμβαστεί με όλε τι πολιτικέ ομάδε και να συμπεριλάβει όλε ε, ή όσο το δυνατόν περισσότερε απαιτήσει. Ε, ωστόσο, η ομάδα μου είναι πολύ δύσκολο να στηρίξει τις εκθέσεις που έχουν να κάνουν με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου, διότι υπάρχουν πολύ καλά σημεία στην έκθεση. Χαίρομαι πάρα πολύ. Αναγνωρίζω εσύ ότι είναι μεγάλη σημασία το να υπάρχει συνέχιση της εδραίωσης επίπεδο του προϋπολογισμού και πρόοδο στι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει. Και εγώ συμφωνώ με τον εισηγητή ότι πρέπει να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα, όχι μόνο με τι συμπίεση του κόστου, αλλά το κόστο θα πρέπει να ανεβαίνει μόνο παράλληλα με την αύξηση τη παραγωγικότητα. Χαίρομαι επίση για αυτά τα οποία αναφέρονται σε σχέση με την απλοποίηση των φορολογικών συστημάτων, για την, ε, επίσης για την ε, απλοποίηση των φορολογικών συστημάτων και τη βελτίωση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης. Από την πλευρά των συντηρητικών περιμένουμε ότι μπορούν να γίνουν ακόμα περισσότερες βελτιώσεις. Αλλά δεν θεωρώ ότι οι οι πολιτικές επιθυμίες που μπορούν να αναφέρουν η ΜΕΝ και οι ΔΕ δεν πρέπει να περιλαμβάνονται σε μια έκθεση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. <clears throat> η συμπλήρωση της νομισματική Ένωσης δεν έχει καμία σχέση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για την ε, οικονομική πολιτική και το συντονισμό. Ο στόχος μας πρέπει να είναι να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα και πάλι θα εκφράσω την αντίρρησή μου με το εργαλείο ανταγωνιστικότητας που ουσιαστικά θέλει να δημιουργήσει ένα αυτόνομο προϋπολογισμό της ζώνης του ευρώ ώστε να γίνει μια ε, οικονομική ζώνη με μεταφορές πιστώσεων. Και επομένως με τις τροπολογίες μου θα αντιμετωπίσω όλα αυτά τα θέματα. Ωραία. Αν θέλει κανείς να πει κάτι πιο διασκεδαστικό, μπορεί. Ο Φίλιπ Λαμπέρς όμως δεν είναι εδώ. Κάπως νιώθω ότι είμαι έκπληκτος γιατί ο Φίλιπ είναι υποχρεωμένος να μην παρίσταται διότι είναι μαζί με την Τρόικα στην Αθήνα, λέει ο Σφεν Γίγολτ, αλλά αιτήσει του έχω ένα βιβλίο για το ιλιουσιν e EL-28 που ήταν ένα αεροπλάνο το οποίο προοριζόταν για να βομβαρδίσει τη Γερμανία κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Θα γυρίσει βέβαια κάποια στιγμή ο κύριος Λάμπερτς. Τούτου λεχθέντος είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένο με την καλή σχέση που είχε και την σωστή μέθοδο με όλου του κοιόδη ηγητέ, μεταξύ των οποίων και τον Φίλιππο Ντεμπάκερ, το αποτέλεσμα το οποίο στο οποίο καταλήξαμε είναι αποδεκτό αποτέλεσμα από τη δική μας πλευρά και μας δίνει θετικά στοιχεία για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο του 2014 και εκτιμούμε ιδιαίτερα την εστίαση που δόθηκε στους στόχους της Ευρώπης 2020 και την ανάγκη να αντιμετωπιστούν υπερβολικές μακροοικονομικές ανισομέρειες μεταξύ των οποίων και υπερβολικό ιδιωτικό χρέος και την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε υπερβολικά πλεονάσματα στο λογαριασμό τρεχουσών συναλλαγών. Μας ικανοποιούν περισσορισμένα μηνύματα τα οποία περιέχονται σε αυτές τις συμβαστικές λύσεις, όπως η αιμονή και η υπογράμμιση της ανάγκης να βελτιώσουμε, να υποστηρίξουμε την κοινοτική μέθοδο και την πρόσκληση προς την Κομισιόν να κάνει μια αξιολόγηση ex post του ρόλου της μέσα στις διάφορες τρόικες. Και να σας πω επίσης ότι η συμπλήρωση της Νομισματικής Ένωσης και η Τραπεζική Ένωση και τα πρόσθετα βήματα είναι, ένα σημαντικό, είναι σημαντικά βήματα μέσα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Δεν βλέπω λοιπόν τις αντιφάσεις αυτές που ανέφερε ο συνάδελφος κύριος Εππινγκ. Ευχαριστώ. Οι ανυποδηματά θα θα εδώ τα 10 λεπτά για να μπορέσει να λάβει το λόγο. Εμείς θα πρέπει να βρούμε κάτι να πούμε τα επόμενα δέκα λεφτά. Δεν έχουμε άλλους σκιώδεις εισηγητές. Εγώ χαίρομαι όπου ο Ήβο μου είπε ότι θα μπορέσει να βοηθήσει να γεμίσουμε τον χαμένο χρόνο. Καλημέρα, Πρόεδρε. Μία σύντομη εξήγηση. θα μπορούσα να πιστέψω ότι ε, ένα αγγλικό βιβλίο θα μπορούσε να γίνει αντικείμενο συζήτηση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Εγώ έζησα ένα τμήμα της ζωής μου από την άλλη μεριά του σιδηρού παραπετάσματος. Και η ψευδέστηση Το Illusion ποτέ δεν βομβάρτισε τη Γερμανία. Για το Illusion πάντως, μου έκανε εντύπωση που ο Φίλιπ Λαμπέρτς γνωρίζει τόσα πολλά, ε, είναι τέτοιο γεράκι, έτσι, τέτοιος πολεμοκάπηλος και έχει μελετήσει και μέχρι και βιβλία για τα βομβαρδιστικά αεροπλάνα. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν, λέει ο Πρόεδρος. Εγώ πήγα σε μια εκλογική περιφέρεια να την επισκεφτώ και επισκέφτηκα μια γεωργική εκμετάλλευση με μια αποθήκη. Στην πραγματικότητα εκεί ε, υπήρχαν ε, τάγκ, τάγκς από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο σε αυτή την, ε, την έκταση. υπήρχαν μικρά βέβαια βρετανικά και μεγάλα γερμανικά. από μινάρια βέβαια, εντάξει. Αλλά σημαντικά. Ε, περιμένουμε την Άννη, προσπαθούμε να γεμίσουμε τον, τον ενδιάμεσο χρόνο. Ίσως με το να θυμόμαστε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν είναι ο καλύτερος τρόπος. Θα μπορούσα να μιλήσω για τις τροπολογίες που έχω υποβάλει. Ε? Καταρχάς, όπως και οι υπόλοιποι, ε, καλωσορίζω το λόγο ύπαρξης αυτού του κανονισμού ε, να διασφαλίσει καλά στατιστικά στοιχεία ε, στα πλαίσια της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών και καλωσορίζω τη δουλειά του εισηγητή, κυρίως στη συμπερίληψη μιας συμφωνίας συνεννόησης για τη συνεργασία μεταξύ της ESS και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όπως και πολλοί άλλοι, οι ειδικέ μου τροπολογίες θέλουν να ενισχύσουν το ρόλο του Κοινοβουλίου στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας και η τροπολογία μου 57 λέει ότι οποιαδήποτε έκθεση της Κομισιόν για παραλήψεις ή για επισκέψεις στα πλαίσια του διαλόγου ε, με βάση το άρθρο 7 πρέπει να υποβληθούν και στο Κοινοβούλιο. Και η 54 επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να επιτρέψουν στα κράτη-μέλη τα οποία ε, είναι υπό εξέταση τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε μία ανταλλαγή απόψεων με την καθήλυνα αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Ένα δεύτερο σημείο το οποίο ε, έχω βάλει στην τροπολογία 45 είναι ότι η διαδικασία θα πρέπει να βασιστεί στην διαδικασία διασφάλισης ποιότητας και να λάβει υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές. Οι προσπάθειες θα πρέπει να πλουστευτούν, ούτως ώστε να μην καταλήξουμε με επικαλύψεις, ε, διπλές προσπάθειες διασφάλισης ποιότητας δηλαδή και παράλληλα στοιχεία. Και ένα τελευταίο σημείο, και εν συνεχεία θα δώσω το λόγο στην Άννη μια και έφτασε, στην ε, τροπολογία 89 θέλω να διασφαλίσω ότι παράγραφος 4 του άρθρου 127 της συνθήκης ε, συμφωνούμε με αυτό και συμμορφωνόμαστε με αυτό ε, όταν, υιοθετούμε, όταν υιοθετούμε, υιοθετούνται συγγνώμη εξουσιοδότηση πράξης. Θα πρέπει να τις καταλάβουμε αυτές και το έβαλα ως υπενθύμηση στην τροπολογία μου. Η Άννη έφτασε και μπορούμε να την ακούσουμε. Ευχαριστώ Σιάρον. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ήμουν στο, σε ένα μποτιλιάρισμα. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για πολλά πράγματα, αλλά δεν ήσουν εδώ, λέει η πρόεδρος. Να ευχαριστήσω και τον Φιλίπ για την εκθεσή του και εν γέννη για την πάρα πολύ επικοδομητική συνεργασία μαζί του <clears throat> που κράτησε σε όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την έκθεση του 2014. Θα κάνω δύο παρατηρήσεις όπως είπα προηγουμένως. Πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα εξισορροπημένη η έκθεση η οποία αντανακλά τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μια κομβική στιγμή λίγους μήνες μόναχα μπροστά από τις ευρωεκλογέ. Για μας ως σοσιαλιστές και δημοκράτες είναι δύο σημαντικά θέματα. Είναι δύο σημαντικά θέματα τα οποία νομίζω ότι ο ΣΥΤΙΣ θα αντιμετώπισε πολύ αποτελεσματικά. Πρώτα απ' όλα το οικονομικό μείγμα πολιτικών και το δεύτερο ο πυλώνας της δημοκρατικής νομιμοποίησης και διακυβέρνησης. Σε ό,τι αφορά την οικονομική πολιτική, καταφέραμε να το κάνουμε σαφές ως κοινοβούλιο ότι η λεγόμενη φιλική δημοσιονομική παγίωση θα πρέπει να είναι η θέση της Κομισιόν έναντι χωρών ακόμα και αυτών που βρίσκονται κάτω από πρόγραμμα προσαρμογής και να περιλαμβάνουν κατευθυντές γραμμές σύγκληση από τη βάση των ψήφισματων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να αντιμετωπιστούν οι μακροοικονομικές ανισομέρειες, όχι στην περίπτωση που υπάρχουν μονάχα ε, ελλείμματα, αλλά και για τις χώρες οι οποίες έχουν πλεονάσματα, να εξασφαλιστεί επίσης υπεραιτέρω ε, δέσμευση για τους στόχους της Ευρώπης 2020 και η ανταγωνιστικότητα αντιμετωπίζεται όχι μόνο ως συμπίεση κόστους, αλλά ως ένα στόχος που μπορεί να επιτευχθεί με τις δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις και με συγκροτημένες προσπάθειες εναντίον της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής καθώς και φοροαπάτης Είχαμε εγκρίνει ένα σχετικό ψήφισμα πριν από λίγου μήνες και ελπίζαμε ότι τουλάχιστον αυτό θα αντανακλάται στην έκθεση αυτή με πιο έντονο τρόπο από ό,τι φαίνεται τώρα και επίσης υπήρχε και μια μνήμα για την καινοτομία, την κοινή αγορά εργασία, την ανάγκη να <clears throat> βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσει να αποκτήσουν χρηματοδότηση. Ό,τι αφορά την οικονομική διακυβέρνηση, νομίζω ότι πετύχαμε να υπάρχει μια σαφής ε, μνήμα για την ε, δημοκρατική νομιμοποίηση στα πλαίσια της οικονομικής διακυβέρνησης και μια σαφέστερη νομιμοποίηση των αποφάσεων που προϋποθέτει μεγαλύτερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μια σαφή μνήμα για την ανάγκη να αντικατασταθεί η λεγόμενη μέθοδος της Τρόικας για τις χώρες που είναι σε πρόγραμμα προσαρμογής με μια ευρωπαϊκού χαρακτήρα <clears throat> νομική ε, οντότητα η οποία θα έχει τα χαρακτηριστικά της λογοδοσίας. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε μια ισορροπημένη έκθεση και θέλω να ευχαριστήσω τον Φίλιπ Ντεμπάκερ για την πάρα πολύ επικοδομητική συνεργασία του και επίσης όλους τους άλλους και όλους Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Τόμας θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να συμμετάσχω στην ε, ε, ομοφροντία επένων που έχει απευθυνθεί στον ε, Φίλιπ Ντεμπάκερ. Παρά το γεγονό ότι δεν έχουμε από του πρασίνου, ο Φίλιπ Λάμπερτ έχει καταθέσει την τοπολογία 13 και θεωρεί ότι ενώπιον των ευρωπαϊκών εκλογών δεν έχουμε κάνει τη σωστή στοχοθεσία για τα θέματα αυτά. Υπάρχει ο φόβος του λαϊκισμού, ο οποίος θα πρέπει να αναχαιριστεί. Εγώ δεν νομίζω ότι ελείπουν αυτά τα στοιχεία στην έκθεση αυτή. Αυτή η έκθεση για μένα είναι πάρα πολύ καλή. Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικέ θέσει από ε, πολιτικέ ομάδε, αλλά οι συγκητέ έχουν καταφέρει να τι συγκεράσουν με ένα θετικό τρόπο. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή είναι ένα καλό μή, μήνυμα. Οι προτεραιότητε λοιπόν οι οποίε είναι πολύ σημαντικέ για όλε τι επιτροπέ μα έχουν λυθεί υπόψη. Είπαμε επίση ότι τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να καταφέρουν να υπάρξουν μέτρα για του προπολογισμού του που θα ευνοήσουν τις μεταρρυθμίσεις, όσο δύσκολες και να απορριφθούν. Επομένως, όλα αυτά δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργήσουν τα ευρωπαϊκά όργανα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και εγώ νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε θετικέ συμβαστικέ λύσει. Έχουμε λοιπόν μια πολύ καλή προσέγγιση. Και θα είναι χρήσιμο να τονίσουμε ότι έχουμε πετύχει μια μεγάλη, ε, ένα μεγάλο αριθμό κοινών θέσεων παρά τις διαφορές μας. Θα είναι απαραίτητο να φανεί και στην προεκλογική εξαρτία ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα, ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συνένεση. Μπορούμε να εμποδίσουμε όλοι μαζί την είσοδο των λαϊκιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αν έχουμε μια τέτοια στεναρική κοινή θέση. Ευχαριστώ. έχουμε χρόνο πάρα πολύ σύντομα στα γερμανικά για να καταλάβει και ο Τόμας. Είναι καλές επιθυμίες και ευσεβείς πόθη που τα σέβομαι όλα αυτά, αλλά η τροπολογία 13 του Φιλίπ δεν αφορά την εργασία που έχει γίνει σε εμά στην Επιτροπή μας, αλλά την έκθεση προόδου της Κομισιόν για την Οικονομική Επισκόπηση. Και εγώ χαίρομαι για τις καλές τροπολογίες των συναδέλφων, αλλά αυτό δεν αφορά την τροπολογία 13. Νομίζω ότι τις καλές ε, επιθυμίες και τους πόθους μπορούμε να τις στείλουμε στη Φραγκφούρτη και να μην τις διεξέλθουμε εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ωραία. Πλησιάζουν οι εκλογές. Ας ξαναδώσω το λόγο στον εισηγητή, στον Φιλίπ. Ε, έτσι είναι. Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους κοιόδης εισηγητές. Ήταν δύσκολο το θέμα και στο παρελθόν να έχει αποδειχθεί ότι αυτές οι συζητήσει πραγματικά δεν είναι εύκολες. Αν δείτε τις τροπολογίες, αν τις έχετε δει, θα καταλάβατε ότι οι θέσεις αρχικά ήταν πολύ διαφορετικές, αλλά τελικά καταφέραμε να φτάσουμε σε μια ισορροπημένη αλλά και δυνατή έκθεση. Δεν έγινε κανένα συμβιβασμό επί της αφήνειας, αλλά στις απόψεις που εκφράζουμε στην έκθεση και στο τμήμα που λέμε για μια δημοσιονομική εξυγίανση φιλική προς την ανάπτυξη, ε, Εκεί έχουμε πει καλά πράγματα. Τα κράτη-μέλη έχουμε πει ότι θα πρέπει να αισθάνονται ότι συμμετέχουν σε αυτή την ιστορία, ότι είναι δική του αυτή η ιστορία, να δείξουν ότι οι αγορέ εργασίες, οι μεταρρυθμίσεις που κάνουν για τα συνταξιδοτικά και για την υγεία, να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να εφαρμοστούν, ε, να τι προωθήσουν αυτέ τι μεταρρυθμίσεις για να πετύχουμε και την ανάπτυξη που θέλουμε. Ευχαριστώ όλου, ευχαριστώ τους κοιόδης συζητητές μου και περιμένω να έχουμε μια θετική ψηφοφορία. Ευχαριστώ, λέει στις 30 Ιανουαρίου ψηφίζουμε, σήμερα δηλαδή, και θα περάσει το θέμα αυτό στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Ευχαριστώ όλους και τον Φιλίπ και τώρα μπορούμε να περάσουμε ε, στο επόμενο σημείο. Είμαστε λίγο νωρίτερα κανονικά, φτάσαμε νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε. Πάμε όμως στο σημείο 4, το οποίο είναι ε, το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας ε, όσον αφορά την τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ. Έκθεση Στρέκερ και θα πρέπει να μας μιλήσει και για τις τροπολογίες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θα μιλήσω για πολεμικά αεροσκάφη. Μπορώ να περάσω στο σημείο μου, το θέμα μου. Ας μιλήσω για κάτι πιο θετικό, που είναι η έκθεση που ετοίμασαμε συνεργασία με τους σκιώδεις ε, εισηγητές. Η πρώτη πρόταση που θα πρέπει να πω θα είναι η έκφραση της εκτίμησης για τη συνεργασία που είχαμε που ήταν πολύ επικοδομητική. Πετύχαμε πολύ καλά αποτελέσματα. Of cooperation, which I am talking about. Μιλώ για αυτό το πνεύμα συνεργασίας, το οποίο φάνηκε όταν συμφωνήσαμε όλοι μαζί σε μια συμβαστική τροπολογία και σε μια προφορική τροπολογία. Ευχαριστώ λοιπόν γι' αυτό όλους τους κοιόδης εισηγητές. Νομίζω ότι έχουμε αρκετό χρόνο. Μπορώ λοιπόν να μακρηγορήσω μπορώ να είμαι χαλαρό. Και πριν ψηφίσουμε για το σημείο αυτό, θα ήθελα να πω ποια είναι τα σημαντικά σημεία τη έκθεση. Τα οποία είναι τουλάχιστον δύο. Το πρώτο. Βασίζεται σε κάτι που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είπε ότι αν γίνει δεκτή αυτή η πρόταση και γίνει και εφαρμοστεί βεβαίως, μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση 50 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μπορούμε δηλαδή να εξοικονομήσουμε έξοδα από το γραφειοκρατικό κόστος, έξοδα που καταβάλουν οι επιχειρήσεις περιτά, όλα αυτά μπορούμε να τα εξοικονομήσουμε. Αυτό είναι το πρώτο, σημαντικό βέβαια. Το δεύτερο, το οποίο θα βρει σύμφωνο όλους που βρίσκονται εδώ. Αυτή η πρόταση μπορεί να βοηθήσει τις διασυνοριακά δραστηριοποιούμενες επιχειρήσεις και να αυξήσει την οικονομική συνεργασία. Όλοι όσοι είχαν να κάνουν ποτέ ε, με ΦΠΑ γιατί είχαν διασυνοριακή δραστηριότητα ξέρουν πολύ καλά ότι χρειάζονται διάφορες απλουστεύσεις, διάφορες προσπάθειες, διάφορα βήματα απλουστεύσεων. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη συνεργασία και τι άλλο να πω. Λοιπόν, από το ΕΛΚ. Κυρία Σάιερ, ευχαριστώ τον εισηγητή μας, ο οποίος πραγματικά δούλεψε πολύ καλά σε αυτό το θέμα. Και όπως είπε, ο στόχος της όλης προσπάθειας είναι να μειώσουμε περαιτέρω το βάρος της επιχειρήσης και να βελτιώσουμε τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Προσπαθούμε να τυποποιήσουμε τις δηλώσεις του ΦΠΑ. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα με, την, με τον κατάλογο ψηφοφορίας εκτός από μία τροπολογία που είναι η τελευταία, η δική μου, η παριθμόν 10, όπου ο εισηγητής τη χωρίζει και έχει βάλει ένα αρνητικό πρόσημο λόγω κάποιων λέξεων. Να σας διευκρινίσω ότι ο στόχος μου δεν ήταν να εξομοιώσουμε τους συντελεστές του ΦΠΑ, να έχουμε έναν δηλαδή συντελεστή, απλώς να δίδονται πληροφορίες με ομοιόμορφο τρόπο. Γιατί αυτό θα ήταν καλό για τις επιχειρήσεις. Αν ξέρουν επιχειρήσεις ότι κάποια πράγματα σημαίνουν αυτό, και υπάρχουν εξηγήσει μονοσήμαντε, είναι πολύ σημαντικό για αυτέ, για να καταλαβαίνουν τι σημαίνουν διάφορα πράγματα και στην άλλη χώρα, στην οποία μπορεί να θέλουν να δραστηριοποιηθούν. Ευχαριστώ λοιπόν για την καλή συνεργασία και είμαι σίγουρη ότι και στο μέλλον θα συνεργαστούμε καλά, ούτω ώστε οι απαιτήσει για το ΦΠΑ και οι πληροφορίε για το ΦΠΑ να είναι τόσο ξεκάθαρε, ούτω ώστε να τι καταλαβαίνουν όλοι. Όλοι οι επιχειρηματίε, όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Ευχαριστώ. Έχουμε σκιώδη ομιλητή ή εισηγητή από τους σοσιαλιστές, δεν νομίζω. Άννη, θέλεις εσύ να μιλήσεις για το ΦΠΑ. Ε, ε, nobody from Aldi speaking, no. Φιλελεύθερη, ο Νίλς δεν είναι εδώ. Ο Σβέν. Εξαφανίστηκε όμως. <laughs> Oh He filled in Philippe and, and has, has um... Ο Φιλίπ δεν χρειάζεται τώρα να αρχίσουμε να μιλάμε για τις ε, αξιώσεις και πάλι. Ήβο. Do you wish to take the floor again? Um... um, um θα θέλεις και πάλι το λόγο. Uh, well, <clears throat> just, uh, just uh, Να καθησυχάσω την κυρία Εσάια. Απολύτως δίκιο έχει. Ο στόχος μου είναι να αποφύγουμε την εναρμόνιση οποιοδήποτε φορολογικού συντελέστη και γι' αυτό ζητάω κατά τμήματα ψηφοφορία και ευχαριστώ για την αιτιολόγηση που δίνετε, την υποστηρίζουμε και τη σεβόμαστε. Μπορούμε έτσι να διευκρινίσουμε τις θέσεις μας. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Και εντάξει, θα έχουμε περισσότερο χρόνο να πιούμε καφέ, δεν πειράζει. Mm. Δίκιο έχετε μου φαίνεται. Έχει προγραμματιστεί ε, για τις 10 παρα 10 η ψηφοφορία και είναι 9 και 40 αυτή τη στιγμή και θα ψηφίσουμε και για αυτό το ζήτημα. Δεκάλεπτο διάλειμμα λοιπόν μπορεί και να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε κάτι για αυτή την τροπολογία σε αυτό το δεκάλεπτο. Πάντοτε είναι μια δυνατότητα. Σε 10 λεπτά, 9 και 50 αρχίζει η ψηφοφορία.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

Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή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

Okay. If you, if you could take your seats. Καθίστε παρακαλώ. thank Είχαμε μια έκτακτη κατάσταση την τελευταία στιγμή, θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα, αλλά πρώτα απ' όλα επανέρχομαι στις ανακοινώσεις της Προέδρου για την ενημέρωση για τους τριλόγους και τα, τη συνέχεια που δόθηκε για τα έγγραφα, για την ε, αποκάλυψη στοιχείων για το TRIPS. Συζητήσαμε λοιπόν όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις αρμοδιότητες των εποπτικών αρχών. Ε, όλα αυτά έγιναν προτού υπάρξει η θέση του Συμβουλίου και τώρα θα γίνει μια προσπάθεια να υπάρξουν Διαπραγματεύσει εν ώψη του επόμενου τριλόγου που θα γίνει στις 18 Φεβρουαρίου. Η άλλη ανακοίνωση που έχω να κάνω είναι ότι υπάρχει μια μικρή διόρθωση στην οδηγία MIFID που έχει διανεμηθεί στα μέλη της Επιτροπής μας <clears throat> χθες 29 Ιανουαρίου και έχει προετοιμαστεί από την ε, Διεύθυνση για τις νομοθετικές πράξεις. Ο στόχος είναι να υπάρξει διόρθωση στο άρθρο 10α μίας παραπομπής, μη φυτένα, μη φυτένα. Βάσει του άρθρου 216 του κανονισμού απουσία οποιασδήποτε αντίρρησης που ήθελε εκφραστεί από την Επιτροπή μας το διορθωτικό θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα ανακοινωθεί στην πρώτη ολομέλεια του Φεβρουαρίου, αν θέλει ο Θεός, και θα θεωρηθεί ότι έχει εγκριθεί εκτός αν υπάρξει μια αντίρρηση από πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον 40 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να ψηφιστεί το διορθωτικό αυτό έγγραφο. Πρόκειται λοιπόν για την ε, παράγραφο 10β4. Επομένως δεν πρόκειται για μια κοσμοϊστορική αλλαγή σε πολιτικές κτλ. Πρέπει επίσης να σας πω ότι ο τρίτος τρίλογος για το SRM έγινε χθε. Συζητήσαμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τις ακάλυπτες πωλήσει την ανάγκη για μια διακυβερνητική συμφωνία, την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας, ε, την ε, σειρά προτεραιότητας των απαιτήσεων των ε, πιστωτών κτλ. Ο επόμενος τρίλογος είναι Τετάρτη στο Στρασβούργο και γίνεται σιγά σιγά πρόοδος, αλλά έχουμε πολλά να πράξουμε ακόμα. Μου ζητήθηκε επίσης να αλλάξω τη σειρά των ψηφοφοριών. Πρώτα το ΦΠΑ λοιπόν. Θα ψηφίσουμε λοιπόν το σημείο 6 πρώτα. Το κοινό σύστημα προστιθέμενης αξίας, φόρ προστιθέμενης αξίας. Μπορούμε να κάνουμε μια ψηφοφορία ελέγχου γιατί ορισμένοι έχουν ξεχάσει τις ε, κάρτες τους. Έχω μονάχα τον debacker. Α, εδώ Τρεις ακόμα δεν έχουν πατήσει το κουμπί τους. 39 είναι στο σύστημα, 37 ψήφισαν. 31 ήταν ικανοποιημένοι, 7 δεν ήταν. Ερχόμαστε λοιπόν στην έκθεση του Ιβο Τροπολογία 4. 4 και 5 μαζί. <clears throat> Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίπτεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 με προφορική τροποποίηση από τον συγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το τελικό κείμενο όπως έχει τροποποιηθεί ηλεκτρονικά Ψηφίσατε όλοι, κλείνω την ψηφοφορία. 39 υπέρ, μία αποχή, καμία ψήφος κατά. Ψηφίζουμε το νομοθετικό ψήφισμα τώρα. Votes Το ίδιο αποτέλεσμα. 39-0 με μία αποχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ, ε, ακούστε με προσοχή. Έχουμε μία ελαφριά σύγκρουση αρμοδιοτήτων επιτροπών για αυτό το ζήτημα. Ε, ήταν σκληρή η μάχη ανάμεσα στη δική μας Επιτροπή και την Επιτροπή Απασχόλησης ε, για το πώς θα το χειριστούμε και τελικά αποφασίστηκε να γίνουν δύο εκθέσεις. Πάντοτε έχουμε πρόβλημα, μπαίνουμε οι ε, μεν στα χωράφια των ΔΕ. και η πρόεδρος ε, της Επιτροπής Απασχόλησης ε, ε, εγκαίρως πριν από δύο μέρες μας ενημέρωσε ότι υπάρχουν δύο προβλήματα. Πρώτον, η, 19, η τροπολογία 19α που αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής Απασχόλησης και συμφωνώ κι εγώ. Δεν μπορώ να το αποκλείσω, αλλά νομίζω ότι οι σοσιαλιστές προτίθενται να αποσύρουν τη 19α όχι, διορθώνει η Πρόεδρος. Είναι η τροπολογία 118 για την ε, παράγραφο 19. Μπορείτε εσείς ε, με χάρη να την αποσύρετε ή εγώ να την κρίνω μη παραδεκτή. Ε, τι λέτε, έχουμε με, τη συμβαστική F, όπου πάλι μπαίνουμε στα χωράφια της Επιτροπής Απασχόλησης, ε, ε, στην Ολομέλεια θα το κάνω θέμα, οπότε για την ε, τη συμβαστική S και όχι F, λέει η Πρόεδρος τώρα. Ένα λεπτό να βρω και τη διατύπωση.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 Ένα λεπτάκι να βρω αυτό που έγραψα πριν από δύο λεπτά και ξαφνικά εξαφανίστηκε μέσα σε όλη τη χαρτούρα όταν έκανα τις ανακοινώσεις μου. Μισό λεπτάκι. Ναι, Άννη, σ' ακούω. Sharon, um, as Πρόεδρε, δεν είχαμε χρόνο. Πέντε λεπτά πριν μα ενημερωθήκαμε για το αίτημα της Επιτροπής Απασχόλησης. Δεν είχαμε χρόνο για να το χειριστούμε δεόντως το ζήτημα. Προτείνουμε ως εκ τούτου να, να τη ψηφίσουμε αυτή την τροπολογία 118 και στη συνέχεια να εξετάσουμε αν πρέπει να την αποσύρουμε πριν από να διεξαχθεί η ψηφοφορία στην Ολομέλεια και για τις ε, τροπολογίες ε, για τη συμβαστική S για να προσθεθεί ε, δηλαδή η αναφορά στο μακροοικονομικό αντίκτυπο της μεταρρύθμισης της αγοράς εργασίας. Αυτό μπορούμε να το δεχτούμε, αλλά και πάλι για την τροπολογία 118 πιστεύω πρέπει να ψηφίσουμε και στη συνέχεια να εξετάσουμε το αν σε μεταγενέστερο στάδιο και πρώτη ψηφοφορία στην Ολομήλεια θα πρέπει να αποσύρουμε την τροπολογία. Πρόεδρος, εγώ δεν θέλω να κάνω αυτό πάλι. Ε, θα την ε, αποκλείσω την τροπολογία 118 εν τη αυτή περίπτωση και δεν θα την ψηφίσουμε για τη συμβαστική ΕΣΕ είτε ε, θα αποκλειστεί είτε στην αρχή που λέμε ότι καλούνται τα κράτη-μέλη να εξυγχρονίσουν την αγορά εργασίας θα πούμε τονίζει, stresses τονίζει το μακροοικονομικό πλεονέκτημα του εξυγχρονισμού από πλευρά των κρατών μελών της αγοράς εργασίας και ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Um, ε, πολύ Πρόεδρε. Ε, συζητήθηκε εκτενώς αυτή η τροπολογία και είναι σημαντικό μας στην έκθεση να δώσουμε έμφαση ε, στις διαστρωτικές μεταρρυθμίσεις αγοράς εργασίας που έχει ιδιαίτερο βάρος, οπότε κατανοώ γιατί τροποποιείται εσεί στη συμβαστική. Οι σκιώδεις ε, ελπίζω να το δεχτούν, αλλά είναι λίγο περίεργο. Εδώ και εβδομάδες τη συζητάμε την τροπολογία και ενημερώθηκα ότι υπήρξε επίσημο σημείωμα της Επιτροπής Απασχόλησης σε σχέση με τον αποκλεισμό αυτών των τροπολογιών ε, για, λόγω σύγκρουση αρμοδιοτήτων. Ο δεν ενημερώθηκε ένα ε, το κρατούμενο, δεύτερον ε, έπρεπε ε, γρηγορότερα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Επιτροπή Απασχόλησης. Προσπαθώ να συνεργαστώ με τον κύριο Γκουτιέρες ούτως ώστε να υπάρχει ισορροπία και μια συνέχεια στην έκθεση, μια συνέπεια και τέθηκαν τα ζήτηματα της αρμο... σύγκρουσης αρμοδιοτήτων. Λοιπόν, και για τις δύο εκθέσεις ε, ε σας ζητώ επίσημα πριν ε, να διεξαχθεί η ψηφοφορία στην Ολομήλεια να κρίνουμε ε, ποια Επιτροπή είναι αρμόδια για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και για την αγορά εργασίας. Πρέπει ξεκάθαρα να δούμε και εμεί στη δική του έκθεση τι έχει μέσα. Αν θέλουν να παίξουν τέτοια παιχνίδια μπορούμε να παίξουμε και εμεί το ίδιο παιχνίδι. Λοιπόν, εγώ θα δεχτώ αυτή την πρόταση αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ περίεργο αυτό ο τρόπο εργασία. Παρακαλώ και εμεί να κοιτάξουμε με ιδιαίτερη προσοχή για να εξετάσουμε το περιεχόμενο της δικής τους έκθεσης, έκθεσης Επιτροπής Απασχόλησης. Πρόεδρος, ναι, ναι, ναι και γι' αυτό σα είπα θα το κάνω θέμα. Στην Ολομέλεια πρέπει να το ε, θέσουμε και στην διάσκεψη των Προέδρων διότι ε, δεν έχουν περισσότερα δικαιώματα και περισσότερες αρμοδιότητες ε, και ε, λυπάμαι που καθυστερήσαμε τόσο πολύ. Ορισμένες φορές είναι δύσκολα τα πράγματα και ως πρόεδρος ε, δυσκολεύομαι καμιά φορά να παρακολουθώ τα πεπραγμένα όλων των υπολείπων επιτροπών. Ε, ε, Φιλίπ, πάντως για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις, γι' αυτό τηρώ αυστηρή στάση και γι' αυτό αποκλείω την τροπολογία 118 και θα ζητήσω από την Πρεβάση να κάνει το ίδιο. Εκείνη είπε ότι υπάρχει μια τροπολογία από την δική της ομάδα γι' αυτό το ζήτημα και γι' αυτό το λόγο αποκλείω την τροπολογία 118 ακριβώς επειδή θα τονίσω τη σημασία του ζητήματος και για τη συμβαστική ΕΣΕ για το μακροοικονομικό αντίκτυπο. Ελπίζω να συμφωνείτε όλοι. Αν τώρα υπάρχουν άλλες προτάσεις για να τροποποιήσουμε περαιτέρω την διατύπωση, θα τις ε, εξετάσουμε στην Ολομέλεια και αν δεν υπάρξει αμοιβαιότητα από πλευρά τη Επιτροπής Απασχόλησης, διότι είναι ίσονος σημασία σε αυτά τα ζητήματα. Βεβαίω τώρα έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω του ζητήματος και μπορεί να προκύψει κλιμάκωση. Θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά πάντως ε, ε, στη διάσκεψη των Πρόεδρων θα το θέσουμε αυτό το ζήτημα. Δεν νομίζω, από όσο μπορώ να κρίνω τώρα, ότι εκείνοι θα αποφασίσουν τελεσίδικα. Ούτω ή άλλω θα τεθεί το ζήτημα στην Ολομέλεια. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στην ε, ψηφοφορία. Έχασα το στυλό μου τώρα. Okay. So, first amendment is amendment. Τροπολογία 13. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές, έλεγχος ηλεκτρονικός, γιατί δυσκολεύομαι σε αυτή την έκθεση. Έλεγχο κάνουμε ηλεκτρονικό. Και στους κατά άλλη μια ψήφο προσθέστε, γιατί εγώ ξέχασα την κάρτα μου. Rejected. Okay. Απορρίπτεται. Ε, συμβαστική α υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβαστική Σ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική D υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική G υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική H υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβασ... τροπολογία 52 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, συμβαστική I υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική J υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική K υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, η τροπολογία 69 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική L υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική M υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική N σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Σε δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 83 υπέρ κατά αποχές δεν είμαι σίγουρη μέσα σε αυτή την αίθουσα τι γίνεται. Επαλήθευση και μην ξεχάσετε να προσθέσετε τη μία κατά. πέρες ψηφοφορίας. Να περίφθη. Συμβαστική ΟΟΥ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Η 88 υπέρ, κατά, η 88 Όχι, 88. Η 87 καλύπτεται από το, τη συμβαστική. Ξεπάμε πάλι. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική π. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 101 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, η R υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αρχικό κείμενο 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 111 υπέρ κατά συγκεκριμένο το αποτέλεσμα. Έλεγχος για την 111, ε, ε, παρακαλώ. Προσθέτουμε ακόμα μία. «20-20 καταπίπτει το αρχικό κείμενο, παράγραφος 18, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβασμός S υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αποκλείσαμε την 118. Ούτως ή άλλως δεν θα περνούσε. Συμβασμός T υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 122 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν ξέρω τι κάνει η ECR. Να το τσεκάρουμε λίγο. Σας τσεκάρω ούτως ή άλλως. Ψηφίζουμε την 122. Ακόμα δύο ψήφους πρέπει να προσθέσουμε. Απορρίπτεται. 124. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 125. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές να τσεκάρουμε το αρχικό κείμενο και προσθέτουμε μία ψήφο υπέρ. Ψηφίζουμε. 21-19 εγκρίνεται λοιπόν. Συμβασμός U, υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβασμός Β, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβασμός W, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 139 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 140 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 141. Με την προφορική τροπολογία των πράσινων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται με την προφορική τροπολογία. Πάμε τώρα στο συμβασμό 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται Συμβασμός Y υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Z, συμβασμός Z υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 2α υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. A, B υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πάμε στις γνωμοδοτήσεις. Παράγραφος 3. Της Επιτροπής Προϋπολογισμών υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 6, budget, υπέρ, κατά. Να το ξανακάνουμε για την 6, παράγραφο 6, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 8, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 9, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 10, υπέρ κατά αποχές μάλλον περνάει. Πάμε τώρα στις αιτιολογικές σκέψεις. Πρώτη τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. δύο. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. τρία. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. τέσσερα. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. AC, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 9, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 10, υπέρ, κατά, τσακάρουμε ηλεκτρονικά το 10. Προσθέτουμε μία ψήφο κατά. Έχουμε 40 άτομα, ε. Εγκρίνεται. Όχι, όχι, λάθος. Καταπίπτει. Καταπίπτει, δεν περνάει. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. AD. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία στο τροποποιημένο κείμενο, παρακαλώ. Προσθέτουμε μία ψήφο υπέρ, τη δική μου. 36 υπέρ, 5 κατά, καμία αποχή. Μπράβο Φιλίπ. Ζητώ συγγνώμη για το θέμα των αρμοδιοτήτων. Και κοίταξε και αυτή την έκθεση, αν θες, που σου είπα. Και τώρα προχωρούμε σε κάτι άλλο, σε κάτι διαφορετικό. Στο σημείο 7 της ημέρας διατάξης. η ενίσχυση της συνεκτικότητας των νομοθετημάτων για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες έκθεση της Επιτροπής μας. Τροπολογία 1 με προφορική τροποποίηση. First of all, paragraphs 1 to 3. Παράγραφοι 1 με 3 συμβούρμπουλες υπέρ. Κατά αποχές δεκτές. Τροπολογία 1 με προφορική τροποποίηση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράφη 5 με 8 το αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 2 με προφορική τροποποίηση της εισηγητρίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράφος 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 με προφορική τροποποίηση της συζήτησης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφοι 12 και 13 το αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 4 με προφορική τροποποίηση, α, με δύο προφορικές τροποποίησεις με την πρώτη προφορική τροποποίηση και τη δεύτερη σαν προσθήκη για να μην υπάρξει σύγκρουση. Λοιπόν, πρώτη προφορική τροποποίηση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τη δεύτερη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφοι 16 και 17 με μια προφορική τροποποίηση υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται το σύνολο με ηλεκτρονική ψηφοφορία Ένα άτομο ακόμα δεν έχει ψηφίσει. Κλείνω την ψηφοφορία. 37 υπέρ, καμία ψήφος κατά και μία αποχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή είναι απλώς μια εκτεσή της Επιτροπής μας, δεν πηγαίνει μετά στην Ολομέλεια. Αυτό είναι για την πληροφόρηση όλων των ενδιαφερομένων και της επερχόμενης Επιτροπής ΕΚΟΝ, της Κομισιόν και περνάμε τώρα στο σημείο της ημέρησης διάταξης υπαριθμών 8. αυτό Okay, we've got one more. Μία ακόμα, ένα ακόμα θέμα στην ημέρηση διάταξη. Μπορείτε να αποχωρήσετε ησύχως και ηρέμος.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 Σημείο 8. Τροπολογίες σε σχέση με το, την έκθεση για τις στατιστικές για την διαδικασία μακροοικονομικών ανισομεριών. Ο εισηγητής είναι ο Dirk Epping. Σας, ευχαριστώ. Όπως υπόθηκε στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων, υποστηρίζω πλήρως το συνολικό στόχο του προτινόμενου κανονισμού για την ε, παροχή και ποιότητα στατιστικών για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Είναι σημαντικό να ενισχύσουμε την μακροοικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα βελτιωμένο στατιστικό σύστημα και σύστημα παρακολούθησης. Βλέπω ότι οι σκιώδεις συγητέ συμφωνούν μαζί μου ότι ο κανονισμός θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί περαιτέρω με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διαδικασίες που προβλέπονται. Και θα πρέπει να εντάσσεται ως ψηφίδα σε ένα μοσαϊκό. Ε, θα πρέπει να υπάρχει, να είναι παράλληλο ε, αυτό που προβλέπετε με το πλαίσιο των μακροοικονομικών, ε, της διαδικασίας μακροοικονομικών ισορροπιών. Ευχαριστώ τους Κιώδης ε, για τη συνεργασία. Την Τρίτη καταφέραμε να συμφωνήσουμε, αν όχι από όλων των σημείων του καονισμού. Οι συμβασμοί που πετύχαμε. Συνοπτικά, πρώτον, διευκρινίσαμε τη διαβίβαση ε, στοιχείων για τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών. Έχουμε μία τελική ημερομηνία μέχρι την οποία η Eurostat μπορεί να συγκεντρώνει ε, στοιχεία για τον πίνακα αποτελεσμάτων του MIP, ούτω ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία διαβίβαση. Μία ημερομηνία επίση ε, δημοσίευση για τα νέα που αναφέρονται στον πίνακα αποτελεσμάτων και δικτών, ούτω ώστε να είναι γνωστά τα αποτελέσματα για λόγου διαφάνεια βέβαια. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το θέμα των λεγόμενων αποστολών και την αποτελεσματικότητα της προκλεπόμενης διαδικασίας. Θέλουμε να μετονομάσουμε τις αποστολές στα κράτη-μέλη ως αποστολές διαλόγου. Είχα προτείνει επισκέψεις διαλόγου, αλλά τελικά συμφωνήσαμε με το αποστολές διαλόγου, για να διευκρινίσουμε ότι είναι μέσα τακτικά ε, ελέγχου. Δεν είναι διεισδυτικά, είναι μια ε, αναθεώρηση ομοτήμων. Τώρα, οι κυρώσεις ε, προκύπτουν μόνο μετά από έρευνα της Κομισιόν για επίτηδε, από πρόθεση παραπίση στοιχείων. Είναι σημαντικό να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στι αποστολέ διαλόγου από τη μία και στις έρευνες από την άλλη, γιατί δεν είναι καθόλου το ίδιο πράγμα. Και τρίτον, θα αντικαταστήσουμε τις ε, εκτελεστικές πράξεις που προτείνει η Κομισιόν με κατεξουσιοδότηση πράξης. Αυτό προτάθηκε από τον κύριο Νουαγκόγκ και υποστηρίχτηκε και από την Επιτροπή ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης με την γνωμοδότησή της. Τέσσερα για τις ε, κυρώσεις, που είναι το βασικό τμήμα του κανονισμού και το πιο επικίνδυνο βέβαια. Σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις για την ε, αλλίωση των στοιχείων, συμφωνήσαμε σε μια διτή προσέγγιση. θα πρέπει καταρχάς, αν χρειαστεί να ε, πληρωθεί πρόστιμο. Το άρθρο 338 της συνθήκης μπορεί να μην επαρκεί ως νομική βάση για την επιβολή κυρώσεων στα κράτη-μέλη. Προτείνω, και το έχω ξαναπροτείνει αυτό, να συμπεριλάβουμε ε, μια τη σκέψη που θα ζητάει από την Κομισιό να εξετάσει την δυνατότητα μια εισαγωγή περαιτέρω νομική βάση, αν χρειαστεί. Και ελπίζω η Κομισιόν να απαντήσει σε αυτό το αίτημα. Φερρυπίν, το άρθρο 121, παράγραφος 6 της συνθήκης, που, συνδέει, που σχετίζεται με την οικονομική διακυβέρνηση, πάνω στο οποίο βασίζεται και η διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών, MIP. Ε, στο πνεύμα συμβιβασμού ε, δεν κράτησα την, τον περιορισμό των κυρώσεων στις χώρες της Ευρωζώνης. Ήταν μια σημαντική παραχώρηση όμως αυτή που έκανα για να φτάσουμε σε συμβιβασμό. Το αποτέλεσμα ποιο είναι, ότι το πλαίσιο για τα στοιχεία MIP δεν θα μπορούν να ταυτίζονται απόλυτα με τη διαδικασία MIP αυτή καθεαυτή, αλλά το επιθυμούν οι άλλοι σκιώδεις συζητητές. Δηλαδή θέλουν οι κυρώσεις να αφορούν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνήσαμε να ευθυγραμμιστεί περαιτέρω το σχέδιο κανονισμού με την ισχύουσα νομοθεσία και τις πρακτικές για τις ευρωπαϊκές στατιστικές. Δεν θέλουμε να επανεφεύρουμε τον τροχό και αν μπορούμε, όπου μπορούμε, να χρησιμοποιούμε ε, την ε, διατύπωση της έκθεσης Μαγκόγκ για τις ευρωπαϊκές στατιστικές. Συμφωνούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τέλος, θα πρέπει να εμπλακεί πιο στενά και πιο νωρί τη διαδικασία και η Επιτροπή μα αυτή, η ΕΚΟΝ, θα πρέπει τη δυνατότητα να ε, καλεί του επικεφαλεί των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών για να συμμετέχουν εθελοντικά σε ακροάσει. Η Κομισιόν θα πρέπει επίση τακτικά να αναφέρεται στο Κοινοβούλιο για την εφαρμογή αυτού του κανονισμού. Ευχαριστώ ακόμα μια φορά τους συναδέλφους για την ε, επικοδομητική συνεργασία σε αυτό το θέμα και ελπίζω να υπάρξει ευρεία συνένεση. Uh, thank you very much uh, for the... Ευχαριστώ. Από το ΕΛΚΑ. Ο κύριος Ντόρφμαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μπορώ να είμαι πάρα πολύ σύντομο. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Έπινγκ ιδιαίτερα για την πάρα πολύ επικοδομητική εργασία του σε αυτό το, σε αυτό το θέμα. Και έχουμε και εμείς παρόμοιες τροπολογίες που θέλαμε να καταθέσουμε, επομένως Είμαστε σε, στην ίδια οδική γραμμή με τον εισηγητή που θα το συναντήσουμε στη συνάντηση των σχεδόν εισηγητών αυτή την εβδομάδα. Και πάλι, χάρη στις ε, προσθήκες που έκανε ο εισηγητής, υπάρχει αυτή η παραπομπή στη διαδικασία MIP Ε, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι οι νέες αυτές διαδικασίες θα συνάδουν με τις προηγούμενες διαδικασίες που έχει δεχθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επομένως η διαδικασία κυρώσεων η οποία έχει εισαχθεί θα πρέπει να συνάδει με αυτά τα οποία δεχτήκαμε στα πλαίσια του Six Και επίσης Θα ήθελα να ισχύουν οι κυρώσεις οι οποίες αναφέρονται εδώ όχι μονάχα στις χώρες της ζώνης του ευρώ αλλά σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω λοιπόν ότι μετά από όλα αυτά μπορούμε να υποστηρίξουμε τη συμβαστική λύση που έχει θέσει ο συγητής με τη μορφή που έχει. Okay, thank you for the... Ευχαριστώ η Άννη για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ, Σάρων, Ευχαριστώ τον Ντίρκ από πλευρά του Λίαμ ε, που ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να παραστεί στη σημερινή τόσο σημαντική συζήτηση. Ξέρετε ότι είναι στην αντιπροσωπεία στην ε, Αθήνα αυτή τη στιγμή, στα πλαίσια τη έκθεση ε, για την έρευνα της ΕΚΟΝ για τη δραστηριότητα της Τρόικα. Ο Λίαμ πιστεύει ότι η συμβαστική που προτείνει η συγκητής που πρότεινε μάλλον πριν από την προηγούμενη σύσκεψη τη Πέμπτη είναι εξαιρετική βάση εργασία. Ω επιτοπλίστων μπορεί να υποστηρίξει αυτέ τι προτάσει και καλωσορίζει το πνεύμα συνεργασία ε, που ε, έχει δημιουργήσει ο εισηγητή. Ο Λίαμ πιστεύει ότι ένα ιδιαίτερα ζήτημα ε, συζητήθηκε διεξοδικότερα αυτή τη βδομάδα. Οι αποστολέ στα κράτη-μέλη μπορεί να υποστηρίξει του συμβασμού στου κατέληξαν οι σκιώδες για αυτό το θέμα. Ο Λίαμ, ωστόσο, θέλει να θέσει ένα ακόμη εκρεμές ζήτημα, αυτό των κυρώσεων. Ο Ντέρκ αναφέρθηκε στις κυρώσεις στα εισαγωγικά του σχόλια σε περίπτωση παραποίησης δεδομένων και στατιστικών στοιχείων. Επί της αρχής ε, προβλέπεται η διαδικασία στον κανονισμό. Ο Λίαμ θέλει να τονίσει ότι το ζήτημα αυτό υπάρχει στο πλαίσιο ε, του κανονισμού πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, ε, για το οποίο θέμα είναι και εισηγητή και προβλέπονται κυρώσεις για όλες τις στατιστικές στοιχείες και σχεδόν με ομοφωνία τον περασμένο Μάρτιο το ενέκρινε η ΕΚΟΝ και στη συνέχεια το Κοινοβούλιο που διαπραγματεύτηκε σε τριμερείς διαλόγους υποστήριξε αυτή τη θέση. Το Συμβούλιο το επέβαλε και στη συνέχεια συμφωνήθηκε ότι το ζήτημα θα το χειριζόμασταν σε τομεακή και σε τομεακά νομοθετήματα, αρχικά στατιστικά στοιχεία για τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπίων, MIP, που συζητούμε σήμερα. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν το αίτημα του Κοινοβουλίου να απηχείται, να αντανακλάται στην τελική έκθεση. Ε, ο Λίαμ πιστεύει επίση ότι το ζήτημα τη νομική βάση μπορεί να λυθεί με το που καταλήξουμε σε πολιτική συμφωνία με το Συμβούλιο για αυτό το ζήτημα και υποστηρίζει την προσέγγιση του εισηγητή για αυτό το ζήτημα. Ευσερχόμενος σε λεπτομέρειες ε, αυτής της συγκεκριμένης διαδικασίας για την επιβολή κυρώσεων, ε, το ΕΛΚΕ προτείνει αντίστοιχες διατάξεις όπως αυτές που υπάρχουν ήδη στη δέσμη 6 οδηγιών. Ε, ρίξει και στοιχείο το οποίο καλωσορίζει ο Λίαμ στη συνέχεια στον κανονισμό επιθυμεί να αναφέρεται συγκεκριμένα δεν πρέπει να εκχωρούνται ε, ε, αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν αυτό δεν είναι απαραίτητο και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εγκαταλείπει το Κοινοβούλιο τις ε, αρμοδιότητες που έχει προς όφελος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γι' αυτό ζητά από τους συναδέλφους της Επιτροπής ΑΕΚΟΝ να υποστηρίξουν τις τροπολογίες 65, 70, 77 έως και 81. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο Σβέν τώρα για τους πράσινους. Και πάλι στο συγγνώμη εξωρώματος του Φιλίππο, ο οποίος είναι στην Αθήνα, μαζί με την ε, αντιπροσωπεία μας για την επίσκεψη σε σχέση με την Τρόικα. Θέλει να ευχαριστήσει τον εισηγητή για την περιεκτική και επικοδομητική προσέγγιση που ακολούθησε μέχρι στιγμής. Καμιά φορά τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συντηρητικού Κόμματο και Μεταρρυθμιστικού ξέρουν πώ λειτουργεί η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορούμε να υποστηρίξουμε σχεδόν όλε τι συμβαστικέ λύσει όπω έχουν, αλλά με μία επιφύλαξη. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε περαιτέρω νομική σαφήνεια σε σχέση με το μηχανισμό επιβολή κυρώσεων που προβλέπεται στο άρθρο 9 και ιδίω σε ό,τι αφορά την ε, συμβατότητά του με την αρχή της ε, αναλογικότητας και τις άλλες πρόνοιες της συνθήκης. Το άρθρο 318 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το αρμόδιο άρθρο. Θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα είχε την δικαιοδοσία για να εφαρμόσει κυρώσεις με χώρες που δεν συμμορφώνονται με αυτόν τον κανονισμό και ιδίως με την υποχρέωση να αποφύγουν θεληματικές παραποίησεις στατιστικών δεδομένων που έχουν να κάνουν με τους δείκτες που είναι η κατάλληλη και η απαραίτητη για την διαδικασία μακροοικονομικών ανισομεριών. Αυτή λοιπόν η διαδικασία που προβλέπεται σε περίπτωση παραβίασης της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος είναι διαφορετική γιατί το άρθρο 258 δεν προβλέπει τη δυνατότητα και το άρθρο 259 τη δυνατότητα να υπάρξει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Υπάρχει επίσης διαφορά από την ε, ε, επίμαχη και οριακή ε, ρύθμιση για κυρώσει τη χώρα στη ζώνη του ευρώ στα πλαίσια τη διαδικασία υπερβολικών ελλημάτων και σε ό,τι αφορά την εφαρμογή δημοσιονομική πειθαρχία στην περιοχή του ευρώ. Και οι δύο αυτέ πρόνοιε βρίσκονται στο εξάπτυχο, το six pack, και βασίζονται στο άρθρο 236 μαζί με το άρθρο 121,6 σε δύο. Και στι δύο αυτέ περιπτώσει ο μηχανισμό κυρώσεων βασίζεται στη δυνατότητα να εγκριθούν περαιτέρω μέτρα τα οποία θα ενισχύσουν το συντονισμό της δημοσιονομικής πειθαρχία όπως προβλέπεται στο άρθρο 136. Και στις δύο περιπτώσεις επίσης, όπως αναφέραμε προηγουμένως, η βάση των κυρώσεων είναι διαφιλονικούμενη μεταξύ των δικηγόρων. Επομένως θεωρούμε ότι το, το δικαστήριο θα μπορούσε να εφαρμόσει χρηματικές κυρώσεις σε κράτη-μέλη που δεν συμμορφώνονται, αλλά δεν θεωρούμε ότι διοικητικού χαρακτήρα ε, χρηματικές ποινές που επιβάλλονται από το Συμβούλιο προτάσεις της Κομισιόν θα ήταν αναλογικό και θα βασίζονται σε μια στερεά νομική βάση. Για αυτό τον λόγο θεωρούμε ότι μια σαφής γνωμοδότηση της νομικής, της νομικής υπηρεσίας μας θα ήταν απαραίτητη πρωτού προχωρήσουμε σε ψηφοφορία για το θέμα αυτό. Ξέρουμε ότι και κάποια μέλη έχουν ε, νομικές επιφυλάξεις για αυτό το λόγο. Αν διατηρηθεί η διαδικασία κυρώσεων και θεωρηθεί ότι συνάδει απόλυτα με την συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να εγκαθιδρυθεί ένα πιο αναλογικό καθεστώς που θα έχει μια πιο βαθμία επιβολή κυρώσεων. Επί τη βάση αυτής της ε, αποδοχής, εμείς θα θέλαμε να έχουμε την ε, αντιμετώπισε δύο στάδια, όπως προβλέπει η τροπολογία 9 που βασίζεται στη δική μας τροπολογία και αυτή του κυρίου Ντόρφμαν από το ΕΛΚ. Αλλά θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια για τη μεταβατική διαδικασία μεταξύ των δύο φάσεων. Καταρχήν θα πρέπει όπως προβλέπετε και στο Six να υπάρξει το κατάλληλο σχέδιο δράση και μόνο σε περίπτωση μη ε, συμμόρφωσης με ένα τέτοιο σχέδιο να επιβληθούν ε, ποινές ως τελική καταφύγη. Σας εύχομαι καλές διαπραγματεύσεις, λέω Φίλιπ. Ευχαριστώ. Έχω υποβάλει και εγώ κάποιες τροπολογίες, δεν χρειάζεται όμως να τις σχολιάσω μια και σχολίασα προηγουμένως όταν μίλησαμε για το εξάμεινο. Για το θέμα της, ε, νομικής, ε, της υπηρεσία. νομικής υπηρεσίας. Δεν έχουμε πολύ χρόνο αλλά μπορούμε να ζητήσουμε από την νομική υπηρεσία της Επιτροπής ΕΚΟΝ, εγκαίρος, πριν την ψηφοφορία. Δεν είναι βέβαια τόσο επίσημη και τόσο πλήρης και δεν προέρχεται από το υψηλότερο επίπεδο της νομικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου, γιατί αυτό θα μας, θα μας έπαιρνε αρκετό χρόνο. Μέχρι να υπογραφεί κτλ. Αν λοιπόν συμφωνείτε, Σβέν, ε, να ζητήσουμε από τη δική μας νομική υπηρεσία της Επιτροπής μας κάνα πρόβλημα. Γίνεται. Ναι, λέει ο Σβέν. Λοιπόν, ο εισηγητή ξανά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να προσθέσω ότι μόλις συμφωνήσουμε για τις συμβαστικές τροπολογίες, θα προσαρμόσουμε τις αιτιολογικές σκέψεις αναλόγως. Οι αιτιολογικές σκέψεις αναφέρονται στο θέμα της νομικής βάσης του κανονισμού. Συμφωνώ ότι η νομική βάση να, είναι πολύ, να μην είναι επακριβώς ευρεία, ε, αρκετά στενή, ειδικά στο διαφορά το θέμα των κυρώσεων. Συμφωνώ λοιπόν εδώ με τον Σβέν. Και θα ήθελα και εγώ να δοθεί νομική συμβουλή από την νομική υπηρεσία. Αλλά νομίζω ότι αρκεί να ζητήσουμε την ε, γνωμοδότηση της δικής μας νομικής υπηρεσίας. Επίσης, ε, θέλω να ρωτήσω την άποψη της Κομισιόν. Την έχω ξαναρωτήσει. Αν η νομική βάση είναι υπερβολικά στενή ειδικά για τις κυρώσει, μήπω θα έπρεπε η παράγραφος 121.6 να συμπεριληφθεί. Αλλά δεν μου έδωσε σαφή απάντηση για αυτό το ερώτημά μου η Κομισιόν. Ελπίζω να υπάρχει εκπρόσωπο τη Κομισιόν εδώ που μπορεί να μα ενημερώσει για αυτό το θέμα. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε το θέμα τη νομική βάση, εάν μπούμε σε διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο. Και θα τεθεί σίγουρα αυτό το θέμα. Ευχαριστώ τον κύριο Ντόρφμαν για τα φιλικά του σχόλια για τις παρατηρήσεις του κύριου Νουανγκόγκ, τι μπορώ να πω, οι κυρώσεις, τα πρόστιμα, συγγνώμη, τα πρόστιμα που υπάρχουν στον κανονισμό είναι το 0,05% του ΑΕΠ. Έφυγε η κυρία Ποδηματά βέβαια, αλλά πρέπει να προσθέσω ότι είναι το ανώτατο όριο δεν επιβάλλεται κατευθείαν αναγκαστικά ένα τέτοιο πρόστιμο το 0,05 του ΑΕΠ. Μπορεί να είναι και πολύ χαμηλότερο το πρόστιμο που θα επιβληθεί. Και να είναι πιο κοντά στα νούμερα που θα ήθελε η κυρία αποδηματά. Επίση έθεσε το θέμα τη νομική βάση και η κυρία Ποδηματά. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να ξεκαθαριστεί και νομίζω ότι η νομική υπηρεσία τη Κομισιόν. Μια και ξέρει, είναι η υπηρεσία γενικά η Κομισιόν είναι το όργανο που ξέρει τα πάντα, θα έπρεπε να μας δώσει ε, στοιχεία. Η διτή προσέγγιση είναι σωστή, είναι ο συμβασμός στον οποίο καταλήξαμε και θα ήθελα να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατό με το θέμα αυτό για να ξεκαθαριστεί η θέση του Κοινοβουλίου πριν το τέλος αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας. Νομίζω τα κάλυψα όλα, δεν ξέχασα τίποτα και χαίρομαι που Αντί για αποστολέ, μιλάμε για αποστολέ διαλόγου. Δεν χρειάζονται ιεραπόστολοι. Οι... Έχουμε εκπρόσωπο της Κομισιόν. Ελπίζω να μπορεί να παρέμβει. Και δεχόμαστε και κραπτές παρατηρήσεις εν συνεχεία μετά τη συνεδρίαση. Κομισιόν. Okay, sometimes they don't work, so... Μερικές φορές δεν δουλεύουν. Αλλάξτε θέση. Ευχαριστώ. Θέλει να τονίσει η Επιτροπή ότι κατά την παρουσίαση της εκθεσής τον Ιούνιο Ελέγξαμε τη νομική βάση, αν το άρθρο 338 δηλαδή επαρκεί για την επιβολή κυρώσεων. Εξακολουθεί να πιστεύει η Επιτροπή ότι το άρθρο 338 είναι επαρκής νομική βάση για αυτό το νομοθέτημα. Ένα σύντομο ερώτημα παρακαλώ, λέει ο Σμεν ε, υπάρχει μια γνωμοδότηση νομικής υπηρεσίας επιτροπής ε, που θα μπορούσατε να μας διαβιβάσετε απάντηση. Γραπτός δεν υπάρχει προς το παρόν. Αλλά ε, για την επιλογή της νομικής βάσης φυσικά έγινε διαβούλευση με την νομική υπηρεσία και επειδή είναι κέρια σημασίας, όταν καταθέσαμε την πρόταση διαβουλευτήκαμε την νομική υπηρεσία. Σφέν Πολλοί θα διασκέδαζαν οι δικηγόροι να το αναφέρουν και γραπτός όλα αυτά και να μας το διαβιβάσετε στη συνέχεια, αλλά σε κάθε περίπτωση θα κάνουμε και μια εξακρίβωση με τη δική μας νομική υπηρεσία, γιατί η μη γραπτή σοφία σας τέθεται να αυτό περιπτώσει, από εμά. Ε, ε, πρόεδρος, ε, καταλαβαίνω την Επιτροπή που λέει ότι όλα τα ελέγχουν, αλλά όταν το Κοινοβούλιο θέτει ένα τέτοιο ζήτημα, λογικό είναι να επανέρχονται και να μας προβάλλουν μια άλλη επιχειρηματολογία για να στηρίξουν ε, τα ε, σημεία που προβάλλουν. Δεν επαρκεί δηλαδή να μας λέτε ότι εσείς το ελέγξατε. Εμείς είπαμε θα αποταθούμε στη δική μας νομική υπηρεσία. Ακούσατε ότι υπάρχουν ανησυχίες. Εάν λοιπόν θα μπορούσατε να μας ε, ε, τεκμηριώστε με κάποιο τρόπο για ποιο λόγο δεν πρέπει να ε, έχουμε τέτοιες ανησυχίες ε, και ότι δεν πρέπει να έχουν ιδιαίτερη σημασία. Να το λάβουμε και αυτό υπόψη. Ευχαρίστω, Γκίγκολτ. Εδώ έχω την γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου, όπου αναφέρει στα συμπεράσματα το άρθρο 9, βάση το οποίο κινείται το Συμβούλιο με τη βάση αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπλα μπλα μπλα. Δεν μπορεί να βασίζεται στο άρθρο 338 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφήστε που έχουν και εμφωλείς για το άρθρο 7. Καλό θα ήταν να επανέλθετε επιτροπή και να σχολιάσετε και αυτό και τη γνωμοδότηση ε, του αδελφού θεσμικού οργάνου. Πρόεδρος, ε, με, στις 12 έχει προβλεφθεί η ψηφοφορία, οπότε ε, είναι ψηλοεπίγη το ζήτημα. Ντέρκ, έχεις τίποτα άλλο να προσθέσεις, είσαι ικανοποιημένος με όλα αυτά. Ωραία. Υποθέτω ότι περιμένουμε τώρα απαντήσεις ε, από τις νομικές υπηρεσίες. Ελπίζουμε να ψηφίσουμε στις 12 Φεβρουαρίου και να πάμε στην Ολομέλεια το Μάρτι. Ε, ίσως χρειαστεί και μια προσαρμογή. Εάν χρειαστεί να επανεξετάσουμε τις ε, γνωμοδοτήσεις των νομικών υπηρεσιών. Ξαναλέω, επίγει το ζήτημα. Θα ε, ζητήσουμε γνωμοδότηση και από τη δική μας νομική υπηρεσία και επίσης εάν μπορούν να έχουν και μια, ένα αντίτυπο τη γνωμοδότηση τη Νομική Υπηρεσία του Συμβουλίου θα βοηθούσε γιατί καλό είναι να ξέρουμε τι πιστεύουν και οι άλλοι. Λίγη και αυτό το θέμα. Η επόμενη μα συνεδρίαση, όπω έλεγα, είναι στις 12 Φεβρουαρίου, 9 και στις 13, πάλι στις 9. Είμαστε στον κύκλο Τετάρτης και Πέμπτης. Απ, έχουμε και το Στρασβούργο την επόμενη εβδομάδα, εκπληξούλα. Οπότε τελικά την Δευτέρα θα, τα ξαναπούμε στην επόμενη συνεδρία.